Καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε τη συνεδρίασή μας. Καλωσορίζοντας την κυρία Τζέιν Λουτζέγκο, που είναι υπουργό ε, Εμπορίου των ε, Ηνωμένων Πολιτειών, αρμόδια για τους ωκεανούς, την ατμόσφαιρα και ε, με βασική αρμοδιότητα το συντονισμό των προσπαθειών για την καταπολέμηση της παράνομης, αδύλωτης και λαθρέας αλίας. Επαναλαμβάνω, καλωσορίζουμε την κυρία Τζέιν Λουστσέγκο. Επαναλαμβάνει ο πρόεδρος, καλωσορίζουμε την κυρία Λουστσέγκο, την Υφυπουργό Οκεανών της των ΗΠΑ και καλωσορίζουμε και την ε, κυρία Δαμανάκη, την Επιτροπό μας που είναι θαμώνα σχεδόν της Επιτροπής και θα της δώσουμε το λόγο για μια σύντομη εισαγωγή. Μετά θα ακούσουμε την κυρία Τζέι Λουστσέγκο και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους συντονιστές πρώτα απ' όλα των πολιτικών ομάδων και στη συνέχεια, όπως πάντα, και με τους βουλευτές που θέλουν να λάβουν μέρος στη συζήτηση. Και φυσικά και η κυρία Λουστσέγκο και η κυρία Επίτροπος, αν επιθυμούν, μπορούν να απαντήσουν. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ για το καλό σωρισμά σας. Αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου. Ήθελα να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που μπορώ να καλωσορίσω εδώ τη δόκτωρα Λουτσάνκο στις Βρυξέλλες και πραγματικά είμαι ευγνώμων στην Επιτροπή Αλίας του Ευρωκοινοβουλίου που διοργάνωσε αυτήν την ακρόαση. Είναι σαφές κατά την άποψή μου, ότι ο αγώνας μας για την βιώσιμη αλία χρειάζεται μια ισχυρή συμμαχία. Γι' αυτό ε, καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να συνεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ. Η Δόκτωρ Λουπτσέγκο είναι από την πλευρά της Αμερικανικής Κυβέρνησης η συνομιλήτριά μου. Είμαι λοιπόν ευγνώμων που προσήλθε σήμερα για να σας δώσει τι πληροφορίες για την ανάλογη πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Ας ξεκινήσουμε από το τι έχουμε κάνει εμείς. Τον περασμένο Σεπτέμβριο υπογράψαμε μια κοινή δήλωση στην Ουάσιγκτον. Το πρώτο βήμα ορόσημο για την ενίσχυση της συνεργασίας μας μεταξύ ε, Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκτοτε έχουμε πάρει και άλλες πρωτοβουλίες. Έχουμε συνεργαστεί για να ενισχύσουμε την καταπολέμηση της παράνομης αλίας και πέραν αυτού έχουμε στηρίξει τα μέτρα συντήρησης και διαχείρισης τα οποία θα επιτρέψουν τη βιώσιμη διαχείριση της αλίας γενικότερα. Από κοινού προσπαθούμε να προσφέρουμε περισσότερη επιστημονική γνώση, καλύτερη συμμόρφωση και ε, περισσότερη προσπάθεια από την πλευρά των αλληλευτικών οργανώσεων. Έτσι, ε, έχουμε ένα νέο ρυθμό στη συνεργασία μας. Ε, στη συνάντηση υψηλού επίπεδου τον Φεβρουάριο επανεπιβεβαιώσαμε την σειρά προτεραιοτήτων μας, ώστε με τη συνεργασία μας να καταπολεμήσουμε περαιτέρω την παράνομη λαθρέα και άναρχη αλληλεία. Και αυτό χάρη στην μεικτή ομάδα Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα ιδρύεται και αρχίζει να λειτουργεί η ομάδα αυτή. Είναι ένα πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν όμω και άλλε εξελίξει στου εννέα μήνε που πέρασαν από την υπογραφή τη κοινή δήλωση. Θα ήθελα να καλωσορίσω ξανά την έκθεση του Κοινοβουλίου για την παράνομη αλεία. Έκθεση που έχουμε πλέον στα χέρια μας ώστε να τονώσουμε μεταξύ άλλων την συνεργασία μας σε ό,τι αφορά τις σημαίες ευκαιρίας ένα από τα βασικά μας ε, προβλήματα. Υπάρχουν πολλά παραθυράκια στο σύστημα, όπως ε, την νιολόγηση ή την αλλαγή σημαία. Αυτά θα πρέπει να πάυσουν, γι' αυτό καλωσορίζω τη σχετική μας απόφαση. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Επιτροπή Αλίας για την αξιόλογη συνεισφορά της σε αυτό τον τομέα. Η παράνομη αλία είναι ένα διεθνές πλέον πρόβλημα, μια ε, ναι, παράνομη δραστηριότητα Οπότε θα πρέπει να κινητοποιηθούν και η Interpol αλλά και η ανάλογη σύμβαση του ΟΗΕ για το διακρατικό οργανωμένο έγκλημα. Και αυτά πρέπει να αξιοποιηθούν στον αγώνα μας και αυτό θα είναι ένα βήμα πρόοδου. Επίσης θα διερευνήσουμε το κατά πόσον μπορούμε να συντονίσουμε τις προσεγγίσεις μας και την οικοδόμηση δυνατοτήτων. Θα πρέπει να ε, ενισχύσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες, τις προσπάθειές τους να συμμορφωθούν με τους ε, διεθνείς κανόνες ε, διαχείρισης. Επίσης, συντονίζουμε τις ενεργειές μας κατά της παράνομης λαθρέας και άναρχης ε, αλίας στην Δυτική Αφρική. Θα ήθελα τώρα να προχωρήσω σε άλλα σημαντικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με την βιωσιμότητα. Τι κάνουμε για τη βιωσιμότητα λοιπόν. Πρώτον, και πριν ε, δώσω τι δικέ μα ιδέε να ποτίσω φόρο τιμής στις Ηνωμένες για, για τα μεγάλα του επιτεύγματα στη διαχείριση των αλλιευμάτων και βάσει των ε, πιο πρόσφατων επιστημονικών πορισμάτων βάσει του νόμου Μάγνουσον Στίβενς. Για να συντομεύω, οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι πιο μπροστά στον αγώνα αυτό σε σχέση με εμά. Μα έχουν ε, δείξει τη σωστή κατεύθυνση για την προστασία τη βιωσιμότητα και μα έχουν εμπνεύσει έχουν ξεκινήσει τέτοιου είδους προσπάθειες πριν από μας, πριν από κάποια χρόνια. Έχω προτείνει λοιπόν τώρα μια πραγματική μεταρρύθμιση της ε, κοινή ε, λευτικής πολιτικής, μια μεταρρύθμιση που πιστεύω ότι θα φέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση στην εμπροστοφυλακή της ε, βιωσιμότητας. Τα μείζωνα προβλήματά μας είναι η απόρριψη και η υπεραλίευση. Θέλουμε λοιπόν να τα αντιμετωπίσουμε. Η καρδιά της δικής μας μεταρρύθμισης είναι να πετύχουμε τα μεγαλύτερα, τα μέγιστα μάλλον αλλιέ. Τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση στο 2015, να αποφύγουμε την υπεραλίευση και να ετοιμάσουμε περισσότερο τις παράκτιες κοινότητες που εξαρτώνται από την αλία. Μέσα από την ε, μεταρρύθμισή μας, τα εισοδήματα των αλλαιών μας και των οικογενειών τους θα αυξηθούν, διότι θα υπάρχουν περισσότερα προϊόντα τα οποία θα εκφορτώνονται. Χρειαζόμαστε μια πιο πράσινη, απλούστερη και τοπικότερη πολιτική. Κάθε δικαίωμα βέβαια, σε κάθε δικαίωμα αντιστοιχεί και μια υποχρέωση. Η ίδια απλή λογική θα πρέπει να ισχύει και για την αλία. Αυτό θέλω να το τονίσω ενώπιόν σας. Εάν λοιπόν θέλουμε να υπάρχουν αλληλευτικά δικαιώματα, εάν θέλουμε να έχουν τέτοια δικαιώματα οι μα, μας, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι και η υγεία των, ε, η ευζοία μάλλον των ε, αλληλευτικών αποθεμάτων είναι κάτι που το λαμβάνουμε υπόψη. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και ελπίζω ότι και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα μας ακολουθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, είμαστε αποφασισμένοι να προωθήσουμε τα ίδια πρότυπα εκτός των ευρωπαϊκών υδάτων, ώστε να ισχύουν σε όλες μας τις συναλλαγές και εμπορικέ εμπορικές σχέσεις, σε όλες τις θάλασσες, ως ε, καλές πρακτικές, ως διεθνής παράγοντας, θα πρέπει να ε, δρούμε υπεύθυνα όπου έχουμε αλληλευτικά συμφέροντα. Στο διεθνές μέτωπο, οι σχέσεις μας με, το, με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ιδιαίτερα πολύτιμες. Συνεργαζόμαστε λοιπόν, αλλά και με, με κυβερνητικές οργανώσεις, με συνομιλητές και εταίρους, με την επιστημονική κοινότητα και με το βιομηχανικό κλάδο, ώστε να καταπολεμήσουμε την παράνομη αλία και να διασφαλίσουμε την βιωσιμότητα. Προκειμένου να είμαστε αποδοτικοί, θα πρέπει να έχουμε τη συμμετοχή όσο των δυνατόν περισσότερων φορέων στον αγώνα μα κατά τη πειρατική αλία. Θα πρέπει λοιπόν να υπογράψουμε σύντομα και μια ακόμη κοινή δήλωση εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ιαπωνία τον Ιούλιο. Αυτό θα είναι το επόμενο βήμα μας. Ελπίζω ότι και άλλοι καθοριστικοί, σημαντικοί μας εταίροι θα ακολουθήσουν σε αυτή την προσπάθεια. Η Δόκτωρ Λουτσένκο και εγώ έχουμε ένα κοινό όραμα και είμαστε αποφασισμένες να συνεργαστούμε στενά βάσει αυτού του πλαισίου. Από κοινού έχουμε περισσότερες πιθανότητες να προωθήσουμε τις αρχές μας και να τις επιβάλλουμε στην αλλήλεια παγκοσμίω. Ελπίζω ότι θα το καταφέρουμε και επίσης ελπίζω ότι η σημερινή συζήτηση εδώ θα επικεντρωθεί ακριβώς σε αυτές τις προτεραιότητες. Ευχαριστώ. Απλ, απλώς, πριν δώσω το λόγο στη Τζέιν, να προσθέσω λίγα λόγια. Θα ήθελα να γνωρίζουν όλοι ότι η Τζέιν είναι πολύ καλή φίλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω όλοι να επωφεληθείτε της παρουσίας της σήμερα, διότι είναι πραγματική τιμή που η δόκτωρ Λουτσέγκο ήρθε σήμερα στις Βρυξέλλες. Σα ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. όντω ε, για όλου μα είναι μεγάλη τιμή και ιδιαίτερα για μένα ω Προέδρο. Έχω την ιδιαίτερη τιμή λοιπόν να δώσω το λόγο στην δόκτωρα Λουτσέγκο. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη τιμή και ευχαριστησή μου που βρίσκομαι εδώ. Αγαπητά μέλη, αγαπητή Επίτροπε, είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση αυτή να έρθω σήμερα είναι τιμή και προνόμιό μου. Ο λόγος που είμαι εδώ σήμερα μπορεί να συνοψιστεί σε τρεις ιδέες που συνδέονται μεταξύ τους. Την ασφάλεια των τροφίμων, την ε, βιωσιμότητα και την οικονομική, το οικονομικό κόστος των τροφίμων. Βιωσιμότητα της αλίας και των υγιών αλλιευμάτων. Πρέπει να δοθεί τέλος στην υπεραλίευση και στην σωστή διαχείριση των ηχθιαποθεμάτων. Είναι κάτι απλό, ωστόσο είναι αρκετά περίπλοκο στην εκτέλεσή του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι δύο από του μεγαλύτερου ε, αλλιευτέ και καταναλωτέ ψαριών και έχουν επενδύσει πολλά. Αυτοί, οι, αυτές οι επενδύσεις μπορούν ε, να δώσουν καρπούς, ε, θέσεις εργασίας δηλαδή. Υπάρχουν πολλά στάδια στην ε, αλλιευτική αλυσίδα, από την παραγωγή, από τους ε, αλληλείς, από, από τους μεταποιητές, από τα εστιατόρια και τους τελικούς καταναλωτές οι θέσεις αυτέ εργασία δημιουργούν ε, σημαντικές ε, προϋποθέσεις για την ευημερία των ε, τοπικών κοινοτήτων. Πάνω από 350.000 άνθρωποι απασχολούνται σε θέσεις εργασίας σχετικέ με την αλληλεία. Έτσι λοιπόν διακυβεύονται πάρα πολλά καθώς εμείς προσπαθούμε να αναθεωρήσουμε το, την ισχύουσα νομοθεσία για την αλληλεία. Γι' αυτό λοιπόν χαιρετίζω και την μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτικής πολιτική. Ε, βλέπω αρκετά κοινά σημεία ανάμεσα στην κοινή αλληλευτική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορούμε να αποφεληθούμε ο ένα από τον άλλο. Και θα ήθελα να σας αναφέρω σύντομα ορισμένα από τα μαθήματα που πήραμε καθώς εφαρμόσαμε τις δικές μας πολιτικές και θα αναφερθώ σε ορισμένες από τις κοινέ μας προσπάθειες. Τα μαθήματα που πήραμε γυρίζουν γύρω από τους εξή τομεί. Καταρχάς, ε, αποφάσεις βασισμένες σε επιστημονική έρευνα, ισχυρή παρακολούθηση και επιβολή των ε, προθεσμιών, περιφερειοποίηση και οι ευκαιρίες που δίδονται στους αλληλείς. Τώρα, η πρόσβαση σε επιστημονική βοήθεια και σε σωστή προσέγγιση είναι ζωτική σημασία για του αλληλεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να τεθεί το ανώτατο όριο αλληλεία σε επίπεδα που θα επιτύχουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Υπάρχει μια γενική συμφωνία, καθώ καταλαβαίνω, στα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη διαχείριση των νύχθη αποθεμάτων για να επιτευχθεί η μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Στι Ηνωμένε Πολιτείε η διαχείριση τη αλεία ελέγχεται από τον νόμο Stevens, ο οποίος ψηφίστηκε πριν από πέντε χρόνια και τέθηκε στα ισχύ το 2006. Η νομοθεσία αυτή, οι ιδιαίτερε τροπολογίε του 2006 έχουν αλλάξει την ε, διαχείριση της αλληλεία στις ΗΠΑ και έδωσαν τα κύρια συστατικά που μας έκαναν πραγματικά ε, ικανούς να αλλάξουμε τα δεδομένα και να επανακτήσουμε τα αποθέματα... σε βιώσιμα επίπεδα. Με το νόμο αυτό του 2006 θέσαμε ανώτατα όρια ε, ψαριάς στα ηχθή αποθέματα βασισμένα σε, επιστημονικές, σε επιστημονικά στοιχεία. Είχαμε περιθώριο 4 ετών για να θέσουμε αυτά τα όρια και να κάνουμε τις έρευνές μας. Πέρυσι το 2011 καταφέραμε να θέσουμε όρια για όλα τα ηχθιαποθέματα που, ελέγχου, που ελέγχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό το επίτευγμα απέτησε τεράστια προσπάθεια. Τώρα όμως έχουμε όλα αυτά τα ανώτατα όρια αλίας. Οι επιστημονικές και στατιστικές επιτροπές μας έδωσαν την αναγκαία επιστημονική καθοδήγηση για να χαράξουμε αυτά τα όρια. Τα υπεραλλιευμένα αποθέματα στις ΗΠΑ... μπόρεσαν να επανέλθουν, να επανακάμψουν και να έρθουν σε επίπεδα μέγιστης βιώσιμης, βιώσιμης απόδοσης. Τα μέτρα αυτά δεν ήταν εύκολο να εφαρμοστούν και υπήρξαν αρκετοί πολέμοι αυτών. Όμως πραγματικά είδαμε ότι επιφέρουν αποτελέσματα χάρη στι ε, θυσίε των αλλιέων και στην νομοθεσία έχουμε δώσει ένα τέλος στην υπεραλίευση. Ένα ψαράς πρόσφατα μου είπε ότι πραγματικά τώρα μπορώ να δω φως στην άκρη του τούνελ. Τώρα έχω μέλλον και αυτό δεν το είχα πριν. Ορισμένα υπεραλλευμένα αποθέματα ε, ανακάμπτουν καλύτερα από κάποια άλλα και επίσης προσπαθούμε να εμποδίσουμε άλλα αποθέματα να υπεραλληλευθούν. Τώρα μερικά σχετικά νούμερα. Μέχρι το τέλος του 2011, 79% των Αμερικανικών ηχθιαποθεμάτων, 174 από τα 288 ηχθιαποθέματα στις ΗΠΑ δεν υπεραλλιεύονται και αλλιεύονται με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. 86% είτε μπορούν να διατηρηθούν από τα, ε, από τα ηχθιαποθέματα τα οποία έχουν υπεραλληλευθεί ε, μπορούν, έχουν δυνατότητα να επανέλθουν. «51 είδη ψαριών βρίσκονται σε διαδικασία ανάκαμψης. Κλειδί σε αυτή τη διαδικασία είναι η αποτελεσματική επιβολή και εφαρμογή των μέτρων αυτών για να σταματήσουν οι παρατυπίες, για να σταματήσει ο αθέμητο ανταγωνισμός και η συνολική αποδοτικότητα τη στρατηγικής μας. Μέχρι τώρα σας ανέφερα ε, επιστημονικές, ε, αποφάσεις που λήφθησαν μετά από επιστημονικές έρευνες, αλλά το κλειδί είναι πραγματικά η περιφερειοποίηση της ε, διαχείρισης της, αλ, οι ίδιοι ε, στόχοι ισχύουν για όλες τις περιοχές, όμως τα επιμέρους ε, τοπικά περιφερειακά συμβούλια αλίας ε, συντάσσουν τα δικά τους σχέδια. Τα σχέδια αυτά πρέπει να εγκριθούν από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και να είναι σύμφωνα με τον νόμο, όμω προέρχονται το καθένα από τι επιμέρου περιοχέ. Διότι αυτέ ξέρουν τι είναι καλύτερο για τα δικά του αποθέματα και καταρτούν ένα μοντέλο κατάλληλο για την εκάστοτε περιοχή. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για την επιτυχία του σχεδίου. Επίσης σημαντικές είναι και οι συζητήσεις που ε, ενθαρρύνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μέρος στη διαδικασία και να, δημιου... και να βρεθούν δημιουργικές λύσεις. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι είναι πιο εύκολο να συμμορφωθούν με, τις, τα νέα δεδομένα και τις απαιτήσει. Και αυτά τα συμβούλια είναι παρόμοια με την μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής εδώ. Μία άλλη πρόκληση στον τομέα της αλληλείας είναι η εναρμόνιση των ε, βραχυπρόθεσμων ερεθισμάτων με, τους, ε, με τα μακρυπρόθεσμα ερεθίσματα. Μέχρι τώρα κυριαρχούν τα βραχυπρόθεσμα συμφέροντα. Όμως μπορούμε να δώσουμε, ε, να δώσουμε σημαντικά ερεθίσματα με τα ακόλουθα εργαλεία για μακροπρόθεσμο συμφέρον. Για παράδειγμα, με τις ε, αλλιευτικές ε, παραχωρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί μεταβιβάζονται άδειες για ε, αλλιευτικές παραχωρήσεις σε αλληλείς οι οποίοι πρέπει να συμμορφώνονται με τα όρια, τα ανώτατα όρια που έχουν δοθεί για το κάθε ψάρι την κάθε χρονιά. Αυτό βελτιώνει την ασφάλεια, βελτιώνει το κέρδος και την ποιότητα ζωής των αλλιέων. Στις Ηνωμένε Πολιτείε, όπου έχει εφαρμοστεί ε, αυτό το σχέδιο έχουμε δει θετικά αποτελέσματα. Εκεί οι αλληλείς δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχούν ή να απειλούνται, διότι μπορούν να, μπορούν να αποφασίσουν οι ίδιοι πότε και πόσα ψάρια θα πιάσουν και σε ποιο, πόσο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν ορισμένε ομοιότητε στα ερωτήματα που ανακύπτουν. Ε, ερωτήματα ολοκλήρωση, ε, οι επιπτώσει ε, στην μικρή κλίμακα. Αυτά που μάθαμε εμεί είναι ότι κανένα από αυτά τα ε, προβλήματα δεν είναι δεν μπορεί να μην αντιμετωπιστεί. Όλα μπορούν να αντιμετωπιστούν. Τα όρια στην ε, ιδιοκτησία και στην ενοποίηση μπορούν να τεθούν. Να τεθούν ε, όρια στο μέγεθος του στόλου, στους λιμένες, σε δανειοδοτικά προγράμματα, τα οποία μπορούν να δοθούν για να βοηθήσουν νέες επιχειρήσεις να εισέλθουν στην αγορά. Περίπου ένα τρίτο των ομοσπονδιακά δικούμενων ε, αποθεμάτων είναι, ε, ρυθμίζονται από αυτά τα προγράμματα, τα, τα catcher programs. Και θα σας δώσω κάποια παραδείγματα για το πόσο ευέλικτο είναι το πρόγραμμα αυτό. Η Αλάσκα έχει ένα από τα πιο προσωδοφόρα θαλάσσια οικοσυστήματα. Δημιουργήθηκε η, ποσόσ... η ποσόστοση το 2004, η οποία επιτρέπει στους ε, κατοίκους της Αλάσκα πρόσβαση στην αλία και επιτρέπει πρόσβαση σε αλείς οι οποίοι δεν είχαν πρόσβαση στα αποθέματα του Βορείου Ατλαντικού και της Δυτικής Αλάσκα. Το πρόγραμμα αυτό είναι ομοσπονδιακό και αφορά 65 παράκτιες μικρές κοινωνίες οι οποίες είναι οργανωμένες σε ομάδες περιφερειακής, ανα... περιφερειακής ανάπτυξης. Εκεί τίθενται ποσοστώσεις για τα ηχθειοποθέματα στον Βερίγκιο Πορθμό και, στα νησιά, και στις Αλεούτιες ε, νήσι. Αυτές οι ομάδες τώρα έχουν αρκετά εκατομμύρια δολάρια κονδύλια να διαθέσουν σε αυτά τα προγράμματα. Μετά, Ορισμένα από αυτά τα προγράμματα έχουν διατάξεις οι οποίες περιορίζουν τις ε, ποσοστώσεις για να διασφαλίσουν ότι η συμμετοχή των ε, μικρών επιχειρήσεων και των ε, κοινοτήτων θα συνεχιστεί. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα για την γλώσσα έχει, έχει περιορισμούς στις ποσοστώσεις και στο μέγεθος του στόλου. Όπως βλέπετε, αυτά τα, τα προγράμματα Catcher είναι μια καλή λύση, δεν είναι όμως πανάκια για όλα τα είδη ψαριών και πρέπει να εξετάζονται κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες της, ε, του κάθε ήχθη αποθέματος. Τα τοπικά και περιφερειακά συμβούλια και τα τοπικά προγράμματα συνεργάζονται με τα Ομοσπονδιακά Συμβούλια για να επιτευχθεί ασφάλεια και στην, ε- στην αλία και στα τρόφιμα. Να περάσω τώρα στην παράνομη λαθρέα και άναρχη αλία. Θέλουμε να σταματήσει η υπεραλίευση και να περάσουμε σε βιώσιμη αηφόρα αλία. Βέβαια έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε, αλλά σίγουρα διαπιστώνουμε ήδη κάποια απτή πρόοδο μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα για την αλία βέβαια θα εξαρτηθεί από την συμμόρφωση όλων με τους κανόνες. Γιατί οι παράνομοι αλίες υπονομεύουν την ασφάλεια των τροφίμων, την, Τα... κέρδη και την νομοτυπία. Η παράνομη πειρατική, η παράνομη λαθρέα άναρχη αλία δυστυχώς σοβεί. Έχουμε τεράστια οικονομική απώλεια μεταξύ και 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο. Η τέτοια παράνομη αλληλεία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αιτία παραγωγής αλληλείας στον κόσμο και ε, υπονομεύει τον αλληλευτικό κλάδο, τους ε, νόμιμους ε, έντιμους αλληλείς και την, τις αλληλευτικές δραστηριότητες. Βέβαια είναι χαμηλού εργασιακού κόστος αυτή η παράνομη αλληλεία γιατί είναι ε, λαθραλής και μάλιστα υπονομεύεται έτσι η προσοδοφορία του ελευτικού κλάδου, καταστρέφονται τα οικοσυστήματα και υπονομεύονται τα ελευτικά αποθέματα. Δυστυχώ, και στον Αμερικανικό ελευτικό ε, στόλο έχουμε εσκεμμένη παραβίαση του νόμου. Εργαζόμαστε σκληρά για να εντοπίσουμε και να διώξουμε τέτοιους λαθραλείς. Επίσης προσπαθούμε να τιμωρήσουμε όλους όσους χρησιμοποιούν ε, εξωαμερικανικές σημαίες ε, για να αλλιεύουν σε αμερικανικά χωρικά ύδατα γιατί υπάρχουν πολλά πλοία με σημαίες ε, που έχουν τέτοιες ε, παράνομες δραστηριότητες αλίας. Χρειάζεται λοιπόν για τον εντοπισμό τους διεθνή συνεργασία. Πέρυσι το Σεπτέμβριο, όπως ανέφερε και η Επίτροπος Δαμανάκη, συνυπογράψαμε μία κοινή δήλωση με διατράνωση το στόχο μας να καταπολεμήσουμε την παράνομη αλία. Και μάλιστα σημειώνουμε πρόοδο προκειμένου να συντονιστούμε και να παρακολουθήσουμε καλύτερα, να ελέγξουμε καλύτερα την ε, εφαρμογή των κανόνων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοστατεί στην αναχέτηση της παράνομης αλίας και θέλουμε να βοηθήσουμε και εμείς την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί πραγματικά η παράνομη αλία είναι ε, η η αρνητική πλευρά της ε, προσπάθειάς μας για η φόρο αλία. Με κοινέ προσπάθειες προωθήσαμε την αθέτηση μέτρων σε περιφερειακά ελευτικά σώματα και σε διεθνή φόρα, προκειμένου να δυσκολεύσουμε τους λαθραλείς να λιεύουν στη θάλασσα, να εκφορτώνουν στα λιμάνια τα προϊόντα τους και να διανέμουν τα προϊόντα τους στις αγορές. Θα συνεχίσουμε να τους κάνουμε τη ζωή δύσκολη με συνεχή επαγρύπνηση. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, ε, βρίσκεται στο πλευρό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσπάθεια πάταξης της παράνομης λαθρείας και άναρχης αελίας. Επίσης, έχουμε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσουμε βιώσιμες ελληνικές πρακτικές παγκοσμίω. Τα τελευταία δύο χρόνια, οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάστηκαν επιτυχώς, προωθώντας προτάσεις για την επιστημονική ε, διαχείριση με βάση την αρχή της προφύλαξης στις περιφερειακές οργανώσεις. Έχουμε αυστηρά μέτρα ελέγχου για τον αριθρό τόνο του Ατλαντικού, Έχουμε ποσοστό που στηρίζονται σε επιστημονικά πορίσματα και προστατεύουμε τα ευάλωτα οικοσυστήματα. Επίσης, απαγορεύεται η εκφόρτωση ευαίσθητων λευτικών ειδών καρχαρία στα λιμάνια. Βέβαια, κάποια είδη καρχαρία ε, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην υπεραλίευση, γιατί είναι αργός ο ρυθμός ανάπτυξής τους, είναι ιδιαίτερα αποδημητικά αυτά τα είδη και τα χαρακτηριστικά αυτών των καρχαριών οδήγησαν σε σοβαρή απειλή του είδους. Η διαχείριση λοιπόν του αποθέματος καρχαρία και η ανάκτηση του ελευτικού αυτού είδους ε, είναι ε, σημαντικό για βιώσιμες λύσεις. Σίγουρα θέλουμε μέτρα βιώσιμης διαχείρισης του, των ειδών καρχαρία και είμαστε υπέρ της πρότασης του ε, Κοινοβουλίου για την απαγόρευση του φίνιγκ και την, γιατί όταν έχουμε φυσική σύνδεση των, των θα βελτιώσουμε και τον τρόπο συλλογής των δεδομένων που έχουμε για τον Καρχαρία. Είχαμε λοιπόν πολύ στενή συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα για ελευθερικά θέματα και προβλήματα. Και ήταν αισθητή η πρόοδος μας μέχρι τώρα. Ακούσαμε για πολύ καιρό ότι θα πρέπει να κάνουμε μια επιλογή μεταξύ περιβάλλοντος και οικονομίας. Όπως γνωρίζετε όμως καλά, αυτή η διχοτόμηση, αυτή η αντιπαράθεση είναι εικονική. Γιατί η υπεραλίευση οδηγεί σε εξαφάνιση των αλευτικών αποθεμάτων και σε εξαφάνιση των ε, αλευτικών θέσεων εργασίας. Μία υγιής οικονομία εξαρτάται από ένα υγιές περιβάλλον. Μπορούμε και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και τα δύο. Η απόφαση για την υφόρο ε, αλία ε, θα εξασφαλίσει κέρδη και για τους αλείς μακροπρόθεσμα και την επιβίωση του κλάδου. Έτσι θα εξασφαλίσουμε και μακροπρόθεσμη επιστημιστική ασφάλεια, θέσει εργασία και οικονομική σταθερότητα για τι παράκτιε κοινότητε. Γιατί σε αυτού του χαλεπού καιρού η επιβίωση τέτοιων ζωνών αποτελεί σημαντική πρόκληση και η απόφαση να, κατα... να καταπολεμήσουμε την παράνομη αλληλεία υποστηρίζει και την, προ... την ανάγκη εξασφάλιση κέρδου και τη βιωσιμότητα. Νομίζω ότι θα πρέπει να δείξουμε θάρρο και διορατικότητα. Αν εγκριθούν οι μεταρρυθμίσει αυτέ, θα απαιτηθούν φυσικά κάποιε θυσίε, αλλά πιστεύω, όπω συνέβη και με τι ΗΠΑ, οι θυσίε αυτέ θα επιβραβευθούν με πολύ μεγαλύτερα ωφέλη. Βέβαια, η δρέψη των καρπών είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Χρειάζεται υπομονή λοιπόν και μακροπρόθεσμη δέσμευση. Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο πλευρό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε αμοιβέ δράσει για να εξασφαλίσουμε τη μακροπρόθεσμη αηφορία τη αλίας που αξίζουν οι συμπολίτε μας. Γιατί η μελλοντική ε, αποτελεσματικότητα του κλάδου ε, είναι κλειδί για την επισητιστική ασφάλεια των επερχόμενων γενεών. Η επισητιστική ασφάλεια, η προσοδοφορία και η βιωσιμότητα είναι αλληλένδετα σημεία που μας ενδιαφέρουν είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και μπορούμε να τα συνδυάσουμε επιτυχώς. Έχουμε βέβαια μακρύ δρόμο μπροστά μας να διανύσουμε για να εξασφαλίσουμε παγκοσμίω ε, ε, βιώσιμη διαχείριση της αλίας. Αλλά η μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής έχουν τον δυναμικό να δημιουργήσουν ένα άλμα πρόοδου προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Muchas gracias, Ωραία, θα περάσουμε τώρα στο γύρο των ερωτήσεων πρώτα των συντονιστών και μετά των υπόλοιπων μελών της Επιτροπής. Θα είναι σύντομος δυστυχώς ο γύρος ερωτήσεων, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ο κύριος Αντινόρο πρώτα, που είναι ο, ε- συντονιστής του ΕΛΚ, ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να καλωσορίσω εξ ονόματος της ομάδας, της ομάδας μου, της ε, ομάδας των το Λαϊκό Κόμμα, ε, την κυρία Λουπτσέγκο. Ήταν διαφωτιστικότατη η παρουσίασή σα. Ευχαριστώ βεβαίω και την Επίτροπο και του συναδέλφου. Ε, ήταν πολύ ενδιαφέρον όσο ακούσαμε. Ε, φίξατε τα σημεία της βιωσιμότητας και της παράνομης αλίας, κυρία Υπουργέ θέματα που μας είναι πολύ σημαντικά και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να εμπνευστούμε από όσα έχετε κάνει εσείς ως τώρα για τη μεταρρύθμιση τη κοινή εκλεκτική πολιτική. Τώρα θέλω να κάνω μια ερώτηση περισσότερο από παρέμβαση. Γιατί θέλω να ακούσω και την άποψή σα για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να βρούμε μια λύση. Βλέπετε ότι η κατάσταση στην Ευρώπη και γεωγραφικώς είναι διαφορετική από ό,τι στι Ηνωμένε Πολιτείε. Η Μεσόγειος είναι μια θάλασσα, θάλασσα περίκλειστη. Και από τις άλλες ε, θάλασσες της Ευρώπης έχει μεγάλες διαφορές. Όμως θα πρέπει να δούμε και τις δικές μας ε, καλές πρακτικές και να σκεφτούμε τι κάνατε και εσείς με τις γειτονικές σας χώρες προκειμένου να σεβαστούν τους κανόνες σας. Παράδειγμα, στη Μεσόγειο, από την Ιταλία από που προέρχομαι εγώ, έχουμε κάποια προβλήματα με τις χώρες της νότιας πλευρά της Μεσογείου. Έχουμε εμεί αυστηρού κανόνες, ε, πολύ συγκεκριμένου για τους αλληλεί μας και τίνουμε να επιβάλλουμε τη συμμόρφωση με αυτού του κανόνες τους αλληλεί μας. Οι όμορε χώρε όμω, ε, η Λιβύη, το Μαρόκο, δεν του σέβονται τους κανόνες αυτούς. Ίσως παρόμοια προβλήματα να είχατε και εσεί με τις γειτονικέ χώρες που όμως δεν έχετε ακριβώς κοινά σύνορα. Ήθελα λοιπόν να μου πείτε κατά πόσον βρήκατε μια λύση σε αυτό το είδο το πρόβλημα. Σε ό,τι μας αφορά είναι αρκετά επιζήμιο. Αυτό είναι μια πρώτη ερώτηση. Αυτή την ερώτηση θέλω να κάνω. Και σε σχέση με τα χωρικά σας ύδατα στον ειρηνικό. Και εμείς πρέπει να σκεφτούμε τι θα κάνουμε με τις χώρες όπου έχουμε κοινά σύνορα και επίσης με την πειρατική αλία. Είναι γνωστό τι κάνουν κάποια πειρατικά σκάφη. Με μια συγκεκριμένη σημαία καταφέρνουν να ε, ξεφεύγουν από τις νομοθετικές δεσμεύσεις. Εδώ έχετε συγκεκριμένη πολιτική που έχετε εφαρμόσει για το θέμα αυτό, συγκεκριμένε τεχνικέ λύσει που θα μπορούσαν και εμάς να μα εμπνεύσουν, να λειτουργήσουν τέλο πάντων ω παράδειγμα και τελευταία ερώτηση για να αφήσω χρόνο και στους υπόλοιπους. Απαριθμίσατε ένα μεγάλο αριθμό αποθεμάτων ειδών όπου επιβάλλατε απαγορεύσεις και σήμερα έχετε πια αποτελέσματα επειδή ακριβώ ε, υπήρξε επαρκή αναπαραγωγή. Ε, λειτουργεί λοιπόν το σύστημα από ό,τι κατάλαβα και με τους αλληλείς που σε τοπικό ε, περιφερειακό επίπεδο εφαρμόζουν την διαχείριση που τους προτείνεται. Όμως, εφόσον υπάρχει ένα μπλοκάρισμα σε κάποια συγκεκριμένα αποθέματα, πώς επιβάλλατε την απαγόρευση στους σε ε, τις περιόδους που είχε πάψει η αλία των συγκεκριμένων ειδών. Μιλάμε για οικονομικούς πόρους που είναι σημαντικοί, γιατί όταν μειώνονται τα εισοδήματα των ελαίων προφανώς τις αρεστώνται σε τέτοιες περίοδους πάυσης. Εδώ Λοιπόν, με ενδιαφέρει κατά πόσον υπάρχουν μέτρα που να μην είναι αντικοινωνικά και θα μπορούσαμε να τα δούμε ω εναλλακτικέ λύσει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Αντινόρο. Παρακαλώ, οι συντονιστές και οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές είναι σύντομοι για να προλάβουν ε, και η κυρία Λουψένκο και η κυρία Επίτροπο ε, να απαντήσουν. Η κυρία Ρόντουστ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και την Επίτροπο και την κυρία Λουτσέγκο. Θα είμαι σύντομη στα ερωτήματά μου. Καθώς καταλαβαίνω, οι Ηνωμένε Πολιτείε κοιτάνε μεγάλο ενδιαφέρον τη μεταρρυθμίσή μας. Θεωρούν την πρόταση της Κομισιόν πολύ θετική. Πώς ορίζετε εσείς τις, ε, την μικρή κλίμακα αλληλεία και την παραδοσιακή αλληλεία Εκεί τι προβλέπετε για την υπεραλίευση επίσης. Είναι αυτά τα θέματα για τα οποία εμείς δεν είμαστε και πολύ σίγουροι. Έπειτα, η περιφερειοποίηση. Πώς λειτουργεί. Ε, μιλήσατε για κάποια αριθμιστικά όργανα, θεωρώ πως εμείς θα τα χρειαζόμαστε. Επίσης χρειαζόμαστε ελέγχους. Πώς ελέγχετε εσείς αν γίνονται παρατυπίες, ε, και όταν αντιλαμβάνεστε ότι έγιναν παρατυπίες, ε, πώς επιβάλλετε κυρώσεις ώστε να αποφεύγονται μελλοντικέ παραβάσεις και πόσα χρήματα επενδύεται στην έρευνα και την καινοτομία. Ευχαριστώ κύριο Στίβενσον. Ο κύριος Γκρο, Γκρομπάρτσικα, δεν κάνω λάθος, ζήτησε το λόγο πριν από μένα. Ναι, συγγνώμη. Κύριε Γκρομπάρτσικ. Δεν σας είδα. Δεν πειράζει κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ε, κύριε Υφυπουργέ, κύριε Επίτροπε. Η ερώτησή μου αφορά το θέμα της περιφερειοποίησης. Μίλησε η κυρία Λουπτσένκο για τις περιφερειακές επιστημονικές ομάδες. Θα μπορούσατε να μας το συγκεκριμενοποιήσετε. Τι μορφή έχουν αυτά τα περιφερειακά επιστημονικά συμβούλια. Συμμετέχουν μόνο επιστήμονες. Ποια είναι η σύνθεσή τους. Ποιος λαμβάνει την απόφαση σε αυτά τα επιστημονικά περιφερειακά συμβούλια. Ποιος συμμετέχει στις συνεδριάσεις συμμετέχουν και εκπρόσωποι των ε, οικολόγων, των συνδικάτων, των αλλιέων ή μήπω ε, σε τέτοιου είδου περιφερειακά συμβούλια συμμετέχουν μόνο επιστήμονες, είναι αμυγό επιστημονικό σώμα. Πριν από ένα μήνα στην Επιτροπή μας οργανώσαμε δημόσια ακρόαση για το θέμα της μεταφοράς λιευτικών ποσοστώσεων, της μεταβίβασης λιευτικών ποσοστώσεων και μάλιστα ο Καθηγητή Μαρσίνκο εκπροσώπησε σε εκείνη τη δημόσια ακρόαση τη ΗΠΑ και μας προειδοποίησε, μα έκρωσε τον κόδωνα του κινδύνου κατά της μεταβίβασης αλληλευτικών ποσοστώσεων. Μάλιστα μας έδωσε ως παράδειγμα την Αλάσκα, ε, η οποία ε, στην οποία ε, εξανεμίστηκε καταστράφηκε σχεδόν πλήρω η αλία μικρή κλίμακα εξαιτία αυτού του συστήματο τη μεταβίβαση των αλληλευτικών ποσοστών. Μπορείτε να μα το σχολιάσετε, παρακαλώ. Κύριε Στίβενσον, εσεί τώρα. Α, συγγνώμη. Αν δεν σηκώνουν το χέρι συντονιστέ, πώ να ξέρω ότι θέλουν το λόγο, κύριε Γκάλεχερ. Ε, να ευχαριστώ ρωτήσω και τους δύο, και την κυρία Λουπτσέγκο και την Επίτροπο που ήρθαν σήμερα εδώ και ευχαριστώ και την ε, κυρία Δαμανάκη που διευκόλυνε αυτήν την ε, συνάντηση. Ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε τις εμπειρίες που είχατε, τις πρακτικές που έχετε εφαρμόσει στις ΗΠΑ σε σχέση με την Αλία και η γλώσσα που χρησιμοποιήσατε, οι όροι, είναι κάτι που καθημερινά ακούμε σε αυτή την Επιτροπή. Επισητιστική ασφάλεια, έλεγχος αλλιευμάτων, βιωσιμότητα, υφορία, κερδοφορία, όλα αυτά, ακόμη και με τα πολιτικά και γεωγραφικά μα σύνορα, δείχνουν ότι έχουμε πολλά κοινά μεταξύ μα. Έχουμε πολλά που θα πρέπει να απασχολήσουν τι σχέσει και τη συνεργασία μα. Πιστεύω κι εγώ, όπω κι εσεί ότι μέλλον υπάρχει αλλά το μέλλον θα υπάρξει μόνο να διασφαλίσουμε ότι η αλία μας είναι βιώσιμη. Ο ψαράς που σας είπε ότι ναι, πιστεύω ότι υπάρχει μέλλον, είναι, εκφράζει μια άποψη που κι άλλοι πολλοί την έχουν εκφράσει. Δεν θα μπορέσει η αλία να επιβιώσει αν δεν υπάρξουν ωφέλη όμως για όλους. Η υπεραλίευση ε, επιδεινώνει την ε, θέση για όλα τα ψάρια και τα αποθέματα, αλλά και με τις τιμές ε, εκφόρτωσης. Για τους καρχαρίες τώρα ήθελα να ρωτήσω. Ε, με αφορμή τους καρχαρίες, τι κάνετε με τις φώκες, τα δέρματα φώκιας που έρχονται από τον Καναδά. Έχω πάει στην Γρινλανδία και ξέρω πολύ καλά τι σημασία έχουν οι φώκες για τον τοπικό πληθυσμό. Ποια είναι λοιπόν η θέση σας για το θέμα αυτό, για τις φώκες, για τις απορρίψεις και πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πολιτική μηδενικής απόρριψης και να έχουμε τελικά κάποια αποθέματα που θα είναι τα αποθέματα του μέλλοντος όσο για την ε, περιφερειοποίηση. Σίγουρα πρέπει να ακολουθήσουμε το νομοθετικό πλαίσιο, όμως μόνο εφόσον ε, ένας τοπικός οργανισμός ε, αναπέμψει κάποιες αποφάσεις σε εσά, λαμβάνονται αποφάσεις στην Ουάσιγκτον. Ή υπάρχουν εκπροσωπήσεις ε, των οργανισμών αυτών. Είναι αυτόνομοι οι οργανισμοί, ανεξάρτητοι. Εκείνοι συνομιλούν με τους διάφορους ενδιαφορομένους στον τομέα ή με εκπροσώπους των αρχών σας. Ευχαριστώ κύριε Λόβεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρους των Πρασίνων θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Λοψέγκο και να πω ότι κάτι που είναι συναρπαστικό είναι ότι εδώ προκύπτει μια πολιτική συνένευση από ό,τι φαίνεται να κρατάμε τα αποθέματα πάνω από το FMSY και να πατάξουμε την υπεραλίευση ενώ το Συμβούλιο φαίνεται ότι το above FMSY θέλει να το καταργήσει, να πει όπου είναι δυνατόν το 2006 πάντως ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε κατάφεραν να εγκρίνουν τον νόμο Μάγνουσον Στίβενς και μάλιστα στη διάρκεια της ε, κυβέρνησης ε, Μπούς και τώρα έχουμε την κυβέρνηση Ομπάμα. Παρ' όλα αυτά συγκεντρώθηκε πολιτική συνένεση. Χρειάζεται πολιτική βούληση για να περάσει ένα τέτοιο νομοθέτημα. Κάτι που λείπει δυστυχώ. Αυτή η πολιτική βούληση λείπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί υπάρχουν ακόμη κάποιε δυνάμει και ε, κάποιε χώρε που είναι επιφυλακτικέ ε, απέναντι στο θέμα αυτό. Οπότε μπορείτε να μας βοηθήσετε, να μας ε, δώσετε κάποιες συμβουλές για να ανακτήσουμε αυτή την πολιτική βούληση. Και Βλέπετε ότι επιτυχάνεται ανάκτηση των ενεχθεί αποθευμάτων, οπότε αρχίζει και καταλαγιάζει και η διαμαρτυρία ίσως που ενδεχομένω δημιουργήθηκε με τον νόμο στους κύκλους των αλλιών. Είπατε επίσης ότι η αλληλεία θα πρέπει να γίνεται κάτω από τα επίπεδα του MSY και με βάση την αρχή της προφύλαξης. Για αυτό το θέμα θα δοθεί μάχη, είμαι βέβαιη, λησαλέα μάχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ο κύριο Γκρομπάρτσικ μίλησε για τα Περιφερειακά Συμβούλια. Άκουσα τόσα θετικά σχόλια για τη λειτουργία των Περιφερειακών Συμβουλίων στι Ηνωμένες που με ενδιαφέρει. Υπήρξε όμω ενδιαφέρον και από Ευρωπαϊκή Πλευρά να έρθουν και να διαπιστώσουν τον τρόπο λειτουργία των Περιφερειακών Συμβουλίων, γιατί φαίνεται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει σύγχυση για το θέμα τη εφαρμογή τη περιφερειοποίηση. Σε ό,τι αφορά τα cut share, στην επιμερισμένη αλία, πιστεύω ότι τέτοιε μεταβάσιμε ε, άδειε δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτικέ, να εναπόκεινται στα κράτη-μέλη. Είμαστε κατά τη ιδιωτικοποίηση των ε, δημοσίων πόρων. Και τέλο, για το θέμα τη παράνομη λαθρέα άναρχης αλίας, χαίρομαι για την προσπάθεια συνεργασία που γίνεται μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ. Οι ΗΠΑ εισάγουν το 86% ε, των ψαριών που καταναλώνουν. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό είναι 60%. Οπότε ε, πώς ε, διαπιστώνετε, πώς εξακριβώνεται ότι τα ελευτικά προϊόντα που εισάγεται είναι νόμιμα ώστε να αποφύγουμε εισαγωγή και τέτοιων προϊόντων παράνομης αλίας. Ωραία. Ολοκληρώσαμε τον κύριο των συντονιστών. Δείξαν το λόγο και τέσσερι ευρωβουλευτέ. Για ένα λεπτό παρακαλώ καθένα, άντε ένα και κάτω, για να προλάβουμε να ακούσουμε και τι απαντήσει. Ο κύριο Στίβενσον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την Επίτροπο Δαμανάκη και την Δόκτωρα Λουτσέγκο. Έχω λίγο χρόνο, αλλά θα ήθελα να κάνω ορισμένε ερωτήσει. Οι Ηνωμένε Πολιτείε λαμβάνουν δημόσια βοήθεια για τον εξυγχρονισμό των σκαφών, των κινητήρων, την κατανα... για να μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων, για την ε, ναυπηγήση νέων ε, πλοίων ή για την διάλυση παλαιών. Υπάρχουν επιχορηγήσεις σε οργανισμούς παραγωγών και αν ναι, για ποιον σκοπό. Επίσης, υπάρχει κάποια βοήθεια στην, ε, όσον αφορά την απόρριψη των ε, ανεπιθύμητων αλλιευμάτων. I hate hearing when the US... Δεν μου αρέσει καθόλου όταν ακούω ότι οι Αμερικανοί τα πάνε καλύτερα από εμά, όμω είστε πηγή έμπνευση. Είναι αλήθεια. Όμω, βλέπετε εδώ σε όλους μας αρέσουν αυτά που έχετε καταφέρει. Προς το παρόν όμως, στο Συμβούλιο και σε αυτήν εδώ την Επιτροπή, στο Κοινοβούλιο, υπάρχουν ακόμα πάρα πολλοί που λένε ότι δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, διότι πρέπει να βάλουμε ε, πρώτα, ε, σε πρώτη προτεραιότητα τους ε, παράκτιους ελίς, τις μικρές κοινότητες, τις δουλειές τους. Αν λοιπόν βάλουμε όρια στη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, θα μείνουν οι άνθρωποι χωρίς δουλειά. Όμως, πραγματικά, εδώ, ε, ο κόσμος ανησυχεί για τι άμεσε επιπτώσει των αλλαγών αυτών και πρέπει να είναι παρόμοια κατάσταση και στις ΗΠΑ. Πολιτείες. Πώς ξεπεράσατε το εμπόδιο αυτό από τις ε, τοπικές κοινωνίες να αλλάξουν μακροπρόθεσμα, αλλά ταυτόχρονα ε, να αποφύγουν τις βραχυπρόθεσμες άσχημες επιπτώσεις. Ευχαριστούμε κύριε Ντέβις. Η κυρία Πατράου Νέβες. Ευχαριστώ πολύ. Σύντομες ερωτήσεις. Πρώτα για τις ε, μεταβιβάσιμες αλληλευτικές παραχωρήσεις. Θα ήθελα να μάθω λίγα περισσότερα για την εμπειρία σας. Σε αυτόν τον τομέα οι ΕΠΑ Πολιτείες τα πάνε πολύ καλύτερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμερίζομαι την άποψη του συναδέλφου. Όμως επιτρέψτε μου να πω ότι αυτά που μας παρουσιάσατε φαίνονται, παρά είναι καλά για να είναι αληθινά και θα ήθελα να μάθω κάποια πράγματα παραπάνω για τα ψηλά γράμματα εάν υπάρχουν, αν δεν υπάρχουν ακόμα καλύτερα. Έπειτα, επίπεδα συγκέντρωση. Όταν λέτε για μεταβιβάσιμε αλλιευτικέ παραχωρήσει, τι εννοείτε και τι απέγινε η αλληλεία μικρής κλίμακας, διότι στη... ήμουν στην Ισλανδία πριν από δύο εβδομάδες και λέγεται ότι η μέθοδος που έχουν για την ε, βιώσιμη διαχείριση είναι πολύ επιτυχημένη. Μετά, άλλο ερώτημα. Ποια υποστήριξη λαμβάνουν οι αλληλείς όσο υλοποιούνται τα σχέδια ανάκαμψης των αποθεμάτων, διότι μας μιλήσατε για την αρετή της υπομονής και για την ανταμοιβή που θα λάβουμε μετά από την υπομονή. Ναι, συμφωνώ ότι θα ανταμοιφθούμε, όμως στο μεταξύ οι ψαράδες και οι οικογένειές τους πρέπει να τραφούν κι αυτοί. Τρίτο ερώτημα, επιστημονική επιστημονικής μελέτης για την ε, διαχείριση. Πώς ε, δουλεύει αυτό το πρόγραμμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, πώς συλλέγεται δεδομένα, για παράδειγμα, πώς ε, χρησιμοποιείται αυτά τα δεδομένα, τι προϋπολογισμό διαθέτεται για την έρευνα πάνω στη θαλάσσια αλία, τι επιστήμονες έχετε, διότι φυσικά είμαι υπέρ μιας ε, βασισμένης σε επιστημονικά στοιχεία προσέγγισης, αλλά πώς θα τη χρηματοδοτήσουμε, εσείς πώς το κάνατε. Και τέλος, μου φαίνεται κάπως ξαφνικό ε, όταν αναφέρατε τους καρχαρίες. Και αυτό το ζήτημα συζητείται ακόμα στο Κοινοβούλιο εδώ για τη μετώπιση των καρχαριών. Δεν ξέρω πώς ε, προέκυψε στην ομιλία σας, αλλά να σας πω ότι πρόσφατα οργανώσαμε ένα εργαστήριο και συνειδητοποίησαμε ότι εάν θέλουμε να συλλέξουμε δεδομένα, ποιοτικά δεδομένα, πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί. Οι αλλοί με εμάς και η πρόταση αυτή ενδεχομένως να, η πρόταση αυτή της Επιτροπής ενδεχομένως να ε, θέσει σε κίνδυνο μια καλή συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα. Ε, Ευχαριστώ. Δύο πολύ σύντομε ερωτήσει. Πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε για την συνάντηση που οργανώθηκε. Πρώτον, η ανάγκη να, υπάρχει, να υπάρχουν προϊόντα λίας είναι όλο και μεγαλύτερη. Τι θα κάνουμε λοιπόν ενώ οι ανάγκε επιστημιστικέ στον πλανήτη αυξάνονται. Θα τους αποδεκατήσουμε τους ανθρώπους. Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν κατά πόσον μια σοβαρή λύση είναι και η ιδιωτοκαλλιέργεια. Και θέλω να ξέρω τι έχετε κάνει σχετικά με το θέμα αυτό στι ΗΠΑ. Το δεύτερο ερώτημα, λίγο πιο ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι το MSY είναι ένα στόχο που θα πρέπει να επιδιώξουμε όσο το δυνατόν συντομότερα. Η μέγιστη βιώσιμη απόδοση αλλά αναρωτιόμαστε αν θα είναι παρκές. Δηλαδή, η θάλασσα μπορεί να είναι ένας τόπος όπου θεωρούμε ότι χωρίς όρια μπορούμε να αλλιεύουμε, αλλά δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της παράνομης αλίας. Υπάρχουν όμως ε, λύσεις πολιτικές ή οποιοδήποτε τύπου ώστε να παράγει περισσότερο η θάλασσα. Δηλαδή τον έχουμε τεράστιες περιοχές όπου δεν επιτρέπεται η αλία για ένα συγκεκριμένο αριθμό ετών. Είναι κάτι που στην πράξη είναι εφικτό, μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνουν τεράστιες τέτοιες προστατευόμενες ζώνες ή αποθέματα που να ε, αυξήσουν την παραγωγή των θαλασσών. Ευχαριστούμε. Ολοκληρώθηκε ο γύρο ε, των ερωτήσεων. Θα δώσω το λόγο στη δόκτωρα Λουψέγκο. Πολλέ ερωτήσει, πληθώρα ερωτήσεων, ελάχιστο χρόνο, αλλά έχω εμπιστοσύνη στην ικανότητα σα να συνοψίσετε αυτέ τι ερωτήσει. Ευχαριστώ για τι καταπληκτικέ σα ερωτήσει. Είμαι βέβαιη ότι δεν θα καταφέρω να απαντήσω σε όλες, αλλά θα επιχειρήσω να απαντήσω τουλάχιστον σε ερωτήσεις που προβληματίζουν τους περισσότερους ευρωβουλευτές. Πολλοί μιλήσατε και ρωτήσατε για την περιφερειοποίηση και πώς λειτουργεί στην πράξη περιφερειοποίηση. Στις Ηνωμένε Πολιτείε, οι 50 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών ε, και μάλιστα όσες ε, έχουν ακτές διαχειρίζουν, τη, διαχειρίζουν την αλία στα παράκτη χωρικά υδάτα μέχρι 3 μίλια από την ακτή. Ανάλογα με την πολιτεία ποικίλει το όριο αυτό. Και η ΝΟΑ, ο δικός μου οργανισμός, είναι αρμόδιος για τα ομοσπονδιακά χωρικά ύδατα, δηλαδή τα τρία μίλια πέραν των 200 ναυτικών μιλίων. Αυτά είναι τα ομοσπονδιακά χωρικά ύδατα. Έχουμε 8 περιφερειακά επιστημονικά συμβούλια διαχείρισης. Νέα Αγγλία, ε, Μέσος Ατλαντικό, Νότιος Καραβι... Καραβική, Δυτική Όχθη, Ειρηνικός, Βόρειος Ειρηνικός, και Χαβάη και τα νησιά του Ειρηνικού. Σε κάθε ένα περιφερειακό επιστημονικό, κάθε ένα από τα περιφερειακά αυτά συμβούλια διαχείρισης ελίας απαρτίζονται από πολλούς εκπροσώπους και εκπροσώπους αλλιέων, επαγγελματιών και ερασιτεχνών, αλλά και άλλους. Ε. Μάλιστα, η διαδικασία σύνθεσης των Περιφερειακών Συμβουλίων περιγράφεται στο νόμο Μάγνουσον Στίβενς θα πρέπει οι άνθρωποι που συμμετέχουν στα περιφερειακά συμβούλια να είναι όχι μόνο αλληλείς, αλλά να είναι και επιστήμονες, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, άλλοι που έχουν όμως γνώσεις περί Είναι ειδικοί για την αλία. Επίση συμμετέχουν εκπρόσωποι και εθνικών και ομοσπονδιακών και πολιτιακών οργανισμών. Κάθε ε, συμβούλιο έχει και μία Επιστημονική και Στατιστική Επιτροπή. Αυτές οι επιτροπές απαρτίζονται αποκλειστικά και μόνο από επιστήμονες που είναι πυρογνώμονε για την περιφερειακή αλία. Ο οργανισμό μας, ο ΝΟΑ, προβαίνει σε αξιολογήσει των αποθεμάτων. Συγκεντρώνουμε δηλαδή δεδομένα για την παρουσία διαφόρων αλληλευτικών ειδών και οι επιστημονικές και στατιστικές επιτροπέ εξετάζουν αυτά τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε εμείς και με βάση τα στοιχεία αυτά και κάποια μοντέλα που εκπονούν υπολογίζουν με ποιο τρόπο και πόσα ε, ψάρια μπορούν να ελευθούν σε κάθε ελευθερικό είδος ανά χρόνο. Και με τις πληροφορίες αυτές ε, δίνονται κάποιες συστάσεις προς το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο είναι η πρόταση που είναι το σώμα που προτείνει ένα ε, σχέδιο διαχείρισης τη αλίας μετά από συμβουλές επιστημονικές. Εμείς το 2006 με τον Μάγνουσο Στίβενς επιτρέψαμε μία από τις σημαντικότερες αλλαγές για τα περιφερειακά συμβούλια. Τα περιφερειακά συμβούλια θα πρέπει να σέβονται τα επιστημονικά πορίσματα δεν μπορούν απλώς να τα συγκεντρώνουν και μετά να κάνουν το κεφάλαιο τους. Θα πρέπει να στηρίζονται σε αυτά τα ε, πορίσματα των επιστημόνων. Και αυτό που προβλέπει ο νόμος Μάγνουσον Στίβενς είναι ε, οι αιτήσει ποσοστώσει ε, και οι άδειε να στηρίζονται σε επιστημονικέ πληροφορίε, να υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση. Επίση, γίνεται έρευνα σε συνεργασία με αλληλεί και πολλά προγράμματα για τη συγκέντρωση στοιχείων για τα ηχθιαποθέματα και για την ε, εξασφάλιση καθαρή αλληλεία χωρίς ε, παραλιεύματα είναι προγράμματα συνεργασία με αλίες. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση λοιπόν χρηματοδοτεί την αγορά ε, των αξιολογήσεων, των εκθέσεων αξιολογήσεων των και έργα των ερευνών ε, που γίνονται σε συνεργασία με τους αλείς. Και με βάση πληροφορίες της Επιστημονικής και της Στατιστικής Επιτροπής, τα Περιφερειακά Συμβούλια προτείνουν ένα σχέδιο διαχείρισης αλίας για κάθε αλλιευτικό είδος ή για ένα σύνολο αλληλευτικών ειδών, όταν πρόκειται για βυθόβια, ας πούμε, είδη. Αυτό το σχέδιο διαχείριση αλληλεία θα πρέπει να εγκριθεί από την ΝΟΑ, το δικό μα οργανισμό. Οπότε χρειάζονται κάποιε κατευθυντήριε γραμμέ ε, που προβλέπονται όμω στο νόμο Μάγκρουσον Στίβεν. Ο επιμερισμό τη αλληλεία, το catch shares, δεν απαιτείται για οποιοδήποτε ελευτικό είδο. Τα επιστημονικά, τα περιφερειακά συμβούλια ε, διαλέγουν την προσφυγή αυτού του μέτρου του επιμερισμού της αλλήλειας ως εργαλείο για τη διαχείριση της αλίας, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Και με αυτό το μηχανισμό χρησιμοποιείται το μέτρο επιμερισμού της αλίας, το cut share. Εμείς ενθαρρύνουμε τα συμβούλια να εξετάσουν την, ε, με την κατανομή των αδειών που χρειάζεται, αλλά ε, τα σχέδια διαχείρισης ε, είναι καρπός διαβούλευσης και διαλόγου σε κάθε, στο εσωτερικό κάθε, κάθε περιφέρειας. Επίσης, οι πληροφορίες για τα χθιαποθέματα, όπως σας είπα, και η έρευνα λαμβάνονται υπόψη στα σχέδια διαχείρισης των περιφερειακών συμβουλίων. Οπότε υπάρχει όντως περιφερειοποίηση. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των περιφερειακών συμβουλίων, γιατί υπάρχουν διαφορές μεταξύ των περιφερειών. Έχουμε ε, περιοχές που είναι πιο κλειστές όπως η Καραϊβική και περιοχές που είναι ανοιχτές όπως ε, γύρω από την Αλάσκα, ο Βόρειος Ατλαντικός. Υπάρχουν διαφορές και ιστορικές και ως προς τη σύνθεσή τους ε, των αλλιευτικών ειδών. Πολύ σημαντική ήταν η ερώτηση της μετάβασης από την υφιστάμενη κατάσταση σε μια πολύ διαφορετική ρύθμιση. Και η ανάγκη είτε οικονομικής είτε χρηματοπιστωτικής ή κοινωνικής προσοχής ή αρρωγής για την διεξαγωγή ε, όσο πιο ανώδυνα γίνεται αυτής της μετάβασης. Αυτό το θέμα είναι πολύ σοβαρό και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν ε, παρακολούθησε τη μετάβαση από την αρχή της, οπότε δεν μπορώ να σας πω για το τι συνέβη στην πρώτη αυτή φάση της μετάβασης. Πάντως πιστεύω ότι σε πολλές περιπτώσεις Υπήρχαν και οικονομικά πακέτα ε, που ενέκρινε το Κογκρέσο για τη μείωση της αλληλευτικής ικανότητας και σε προγράμματα που ίσχυσε ο πλημμυρισμός αλληλείας, το Card δεν έγινε κάτι τέτοιο. Είναι, ισχύσε ένας ε, μηχανισμός αγοράς για την δυνητική μείωση της αλληλευτικής ικανότητας, ώστε να μπορούν οι που για παράδειγμα δεν έχουν και πολύ καλές ε, επιδόσεις να εξαγοραστούν από άλλους. Είναι ένας από τους μηχανισμούς ε, οι παραχωρήσεις, αυτό το cut share. Δεν είναι υποχρεωτική όμως η εφαρμογή τους. Ε, στις πρώτες μέρες εφαρμογής των προγραμμάτων cut share δεν υπήρχαν έλεγχοι, ε, στην, δεν υπήρχαν αρκετοί έλεγχοι και έτσι έγινε μια ενοποίηση και σίγουρα εκεί η αλληλείς μικρή κλίμακο ήταν αυτή που βγήκαν χαμένοι στην πρώτη φάση εφαρμογής του συστήματος του cut Shares. Και φαίνεται ότι ήταν προβληματικό αυτό το σύστημα για κάποιες κοινότητες και για τα μικρά σκάφη. Με βάση την εμπειρία αυτή, έχουμε συνδέσει νέα προγράμματα επιμερισμού των αδειών, ώστε να αποφευθεί εξόντωση των αλλιών μικρής κλίμακας. Οπότε ένα πρόγραμμα ε, cut share μπορεί να δομηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε ένα τμήμα των ποσοστώσεων να, να ε, αφιερώνεται σε συγκεκριμένη κοινότητα, να κρατείται για συγκεκριμένο μέγεθος αλλιευτικών σκαφών, ώστε να προστατευτούν οι μικρές κοινότητες και οι μικρής κλίμακας αλλιείς. Μην θεωρείτε λοιπόν ότι οι παραχωρήσεις αυτές κατά ανάγκη έχουν αρνητικές επιπτώσεις. Το κάτσερι έχει κατά ανάγκη αρνητικές επιπτώσεις. Απλώς υπάρχει τέτοια δυνατότητα, ε, μερικές φορές οι λεπτομέρειες κρύβεται ο σατανάς όπως λέμε. Προσπαθούμε να δαχθούμε από τα παλιά παθήματα και τα νέα συστήματα, τα νέα προγράμματα cut-share, παραχωρήσεων προσπαθούν να αποφύγουν τις αρνητικές συνέπειες που εντοπίσαμε στο παρελθόν. Δεν ξέρω, ίσως εξάντλησα το χρόνο μου. Ανέφερα λοιπόν ότι το θέμα των παραχωρήσεων των cut shares προτείνεται από το Συμβούλιο, από τα Περιφερειακά Συμβούλια. Δεν είναι κάτι που προτείνεται σε κεντρικό ομοσπονδιακό επίπεδο. Η προσέγγιση μας ως προς τις απορρίψεις Ε, επενδύει σε κοινή έρευνα, σε συνεργασία με τους αλείς, ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο η παραλίευση, η παρεμπίπτουσα αλία, με τη χρήση επιλεκτικών ε, δικτύων, ή με συσκευές ώστε να αποφεύγεται η εμπλοκή και χελωνών στα δίχτυα και ούτω καθεξής. Επίσης, κάτι άλλο που ανακαλύπτουμε με το σύστημα cut shares, με τις παραχωρήσεις αυτές, είναι ότι δίνονται ενάψματα στους αλείς να περιορίσουν στο ελάχιστο την παρεμπίπτουσα αλεία. Και αν όντως μπορούν να υποφεληθούν από αυτόν τον περιορισμό της παραλίευσης, σε πολλά προγράμματα cut shares, ε, βλέπουμε ότι οι απορρίψεις έχουν ε, μειωθεί αισθητά, γιατί οι αλληλείς είναι πολύ έξυπνοι και ξέρουν πού να ψαρεύουν και ξέρουμε τι τρόπο να ψαρεύουν, ώστε να ελαχιστοποιήσουν την αλίευση ανεπιθύμητων ειδών και να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους. Οπότε, σε προγράμματα τέτοιων παραχωρήσεων, cut shares, διαπιστώνουμε πολύ αισθητή μείωση των ανεπιθύμητων αλλιευμάτων της παρεμπίπτουσας αλλίας. Και μάλιστα στην Καλιφόρνια έχουμε ένα νέο πρόγραμμα cut share, που υιοθετήθηκε τον Ιανουάριο του 2011 για ένα πολύ πλούσιο σύμπλεγμα βυθόβιων ειδών και μερικά τέτοια βυθόβια είδη είναι πολύ σπάνια. Με αν αλλιεύονται πολλά τέτοια σπάνια βυθόβια είδη, τότε η αλία για τον κάτοχο της ποσόστοσης εξαντλείται για τον δικαιούχο. Είναι πολύ σημαντικό αντικίνητρο για να αποφευθεί η αλλίευση σπάνιων ειδών. Οπότε αυτό που κάνει ο αλίας είναι να συγκεντρώνει ε, κάποιες πληροφορίες και να συνεργάζεται με άλλους ε, αλληλείς, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος αλλήλευσης τέτοιων ε, ε, σπάνιων ειδών. Στην ανταλλαγή λοιπόν των πληροφοριών, με πολύ έξυπνο τρόπο προσπαθούν οι αλληλείς να αποφεύγουν τα ανεπιθυμητά είδη και να επικεντρώνονται στα κερδοφόρα. Και πραγματικά μέσα σε ένα χρόνο μετά την εφαρμογή αυτού του συστήματος έχουν εξακοντιστεί στα ύψη τα κέρδη των αλλιών. Το θέμα της πολιτικής βούλησης είναι επίσης πολύ σημαντικό. Ε, ο νόμος Μάγνουσον Στίβενς ε, πρωτοπέρασε το 1975. Ε, είχε μεγάλη υποστήριξη γιατί υπήρχε έντονο φαινόμενο υπεραλίευσης. Ήταν καλός αυτός ο αρχικός νόμος, καλοπροαίρετος, αλλά δεν είχε την αυστηρότητα ως προς τα χρονοδιαγράμματα, την παρακολούθηση, τα, τις πως ποσοστώσεις για κάθε ελευτικό είδος, δεν είχε ε, τις δυναμικές και αυστηρές τροπολογίες που είχε ο νόμος του 2006. Και όλα αυτά τα σημαντικά σημεία του νόμου του 2006 οδήγησαν σε ε, μεγάλη ε, υποστήριξη του νόμου και μία πρωτοπορία των βασικών επιτροπών που συγκέντρωσαν τα διάφορα τμήματα της νομοθεσίας, ε, ε, τα ομοδοποίησαν και κατέθεσαν την νομοθετική πρόταση Μάγνουσον Στίβες παρά κάποιες έντονες διαμαρτυρίες και παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισαν ε, οι ελληνικές κοινότητες. Ήταν δύσκολη η πορεία, πάντως θα πρέπει να έχουμε κατά νου το μέλλον να έχουμε μια διορατικότητα και να λαμβάνουμε σήμερα κάποιες σωστές αποφάσεις, ε, ε, λαμβάνοντας υπόψη όμως τον μελλοντικό ορίζοντα και το θέμα της μετάβασης. Να δούμε τι συνέπειες θα έχει η μετάβαση, ποιες είναι οι κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες ε, που θα προκύψουν από τη μετάβαση και πώς μπορούν να μετριαστούν. Μερικοί που στις Ηνωμένε Πολιτείες βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα της μετάβασης ίσως έχουν πολύ περισσότερα να σας πούν. Πάντως ε, θεωρώ ότι αναφυσβήτητα δρέπουμε σήμερα τους καρπούς ε, λίγα χρόνια μετά της σοφίας και της πολιτικής βούλησης των ε, πρωτοπόρων του νόμου Μάγνουσον Στίβενς. Είπατε ότι φαίνονται τέτοιες ιστορίες που σας περιγράφω ιδε, ιδεώδεις, ιδανικές για να είναι αληθινές. Δεν ήταν ανώδυνη η πορεία μας αλλά βλέπουμε επιτέλους ε, τα πλεονεκτήματα μιας ισχυρής και αυστηρής ομοθεσίας. Το περιφερειακό σχέλο, η αρχή της προφύλαξης, όλα αυτά συνδυάζονται στο νομοθέτημα αυτό και μας φέρουν σε μια πολύ καλύτερη θέση σήμερα από ό,τι στο παρελθόν. Πιστεύω ότι μπορούμε, να διδαχθούμε ο ένας από τον άλλον, να διδαχθούμε και από τα παθήματά μας, να αξιοποιήσουμε τις ε, καλές γνώσεις και πρακτικές για να έχουμε υγιείς ωκεανούς, επιστηστική ασφάλεια, βιωσιμότητα της αλίας. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Το θέμα είναι πώς θα τα υλοποιήσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Λουπτσέγκο, δόκτωρα Λουπτσέγκο. Οπότε ολοκληρώνουμε αυτό το σκέλος της συνεδρίασης. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Ξέρετε ότι οι πόρτες της Επιτροπής μας είναι ανοιχτά, ε, ανοιχτές διάπλατα και για σας και για την κυρία Επιτροπό φυσικά. Σας αποχαιρετούμε και συνεχίζουμε και κλεισμένο το θηρό για το επόμενο θέμα.